Μας λείπει ακόμη μία ψήφος. Πέρας. Ψηφίσατε όλοι. 33 υπέρ, 2 κατά, 0 αποχές. Κυρία της Άλντε, έχετε την κάρτα σας. Α, πολύ ωραία. Οπότε εγκρίνεται και συγχαίρουμε τον εισηγητή μας. Και τώρα, να ψηφίσουμε την έκθεση Σαλβαδόρ Γαρίγα για την Λομβαρδία. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Έχουμε 7 τροπολογίε του συναδέλφου Νταρντέν. Να τι ψηφίσουμε μαζί. Όχι. Καλά. Ο εισηγητή βέβαια είναι υπέρ. Όχι, ο εισηγητή είναι υπέρ όλων. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά η φιλελεύθερη 8, 9 αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά ένας κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά Δύο ψήφοι κατά. Αποχές εγκρίνει. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Δύο ψήφοι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Δύο ψήφοι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα στην τροπολογία 8 έχουμε μια προφορική τροπολογία τη οποία έχετε το κείμενο υπέρ. Κατά. 8 αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 9 των φιλελευθέρων, ο εισηγητής είναι κατά. Αλλά καταπίπτει, διότι εγκρίθηκε η 8, έτσι δεν είναι. Ωραία, τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική παρακαλώ. Άρχεται. Λείπει μία ψήφος. Παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρας. 33 ε, κατά εγκρίνεται. 2 κατά εγκρίνεται. Να περάσουμε τώρα στην ε, ψήφιση της εκθέσεως ε, της Κατρίν Τροτμάν για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τρεις τροπολογίες της από κοινού. Ωραία, υπέρ, παρακαλώ. Κατά Τέσσερις κατά εγκρίνονται. Τροπολογία 5 που προτείνει μια νέα παράγραφο της κυρίας Καρβάλιο. Α, με συγχωρείτε. Α, με Α, δεν είδα την 4. Η τροπολογία 4, Καρβάλιο, υπέρ. Και ο συγκητής βέβαια είναι υπέρ. Κατά. Μία ψήφος κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, 5 με την προφορική τροπολογία που θα πρέπει να έχει στόχο τη σωστή αντιμετώπιση υπέρ, κατά, αποχές, ωραία, τρεις κατά αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Πέρας, ψηφίσατε όλοι, ωραία. 33 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Ίδιος σχετισμός. Συγχα... Συγχαίρουμε την κυρία Καθρίν Χοτμάν έκθεση Έιντερ Γκαρδία Θάβαλ. Δεν θα σας διαβάσω τον τίτλο γιατί ε, θα κρατήσει πιο πολύ την ψηφοφορία. Λοιπόν, να ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες 7, 2 και 5 που συμπίπτουν. Η συγκίτρια είναι κατά γιατί τις έκανε ίδια υπέρ, κατά, Ωραία, θα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, γιατί υπάρχουν αρκετές ψήφοι κατά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 23 υπέρ, 13 κατά. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Τροπολογία 8. Έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Να καταργηθεί η φράση αυτή που λέγεται τα κράτη-μέλη των οποίων η πολιτική συνοχή κτλ. υπέρ κατά δώδεκα κατά αποχές ίδιος σχετισμός ωραία δεύτερο τμήμα να ψηφίσουμε για την παράταση 2011 έως 2013 υπέρ κατά Οκτώ αποχές εγκρίνεται επίσης. Ε, λίγο διαφορετικός σχετισμός. Εννέα της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Επτά κατά αποχές. Είστε υπέρ κατά παρακαλώ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Μάλιστα. Και η Έλγα υπέρ. Λοιπόν, υπέρ ποιοι είναι παρακαλώ. Τροπολογία 9. Ωραία. Κατά. Ωραία, αποχές, καλά. Ε, ε, εγκρίνεται. Στον τίτλο τώρα. Τροπολογία 1 Τι ηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Ωραία, εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 3 της συγκίτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 της Γκουε. Είναι συμβατή με την 3. Η συγκίτρια είναι υπέρ, υπέρ. Παρακαλώ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Τέσσερα της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έντεκα της Γκουε. όπως προηγουμένως είναι συμβατή συγκίδρια υπέρ. Υπέρ παρακαλώ οι έντερ και οι σοσιαλιστές και η Γκουε. Κατά. Οι περισσότεροι απορρίπτεται. 6 της εισηγήτριας. Α, να μην την ψηφίσουμε. Καλά, ωραία. ωραία. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. 37, 37 περισσεύει. Καλά. Κάποιο ε, ε, εισήγαγε την κάρτα του, αλλά την έβγαλε αμέσω. Εμπάσχετο. Πέρα. 26-8-2. Εγκρίνεται. Τελευταία ψηφοφορία. Έκθεση Utah Haug. Τροποποίηση του κανονισμού για την, τον οργανισμό GNSS. Συμφωνούμε όλοι να ψηφίσουμε από κοινού τις τροπολογίες. Ωραία, μία μόνο ψηφοφορία. Και τελική και επί των τροπολογιών. Ωραία, ηλεκτρονική τότε. Η ηλεκτρονική. Και για τι τροπολογίε όλε και για την τελική έκθεση. Γιούτα είναι όλα ή τίποτα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πέντε ψήφοι υπέρ και μία κατά. Κάποιος είναι μπαγάσας. Και μηδέν αποχές. Ναι, αλλά αυτή η μία ψήφος κατά ε, διαφυλάτει την ε, ε, διαφορετικότητα στην, στο όργανό μας. Αλλιώς θα ήμασταν στα Τελειώσαμε τις ψήφους, τις ψηφοφορίες. Επί των εκθέσεων πρέπει να ψηφίσουμε ορισμένες μεταφορές πιστώσεων. Μήμα 3 του 2013 το ΕΛΚ μου είπε ότι κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Τζοβάνι Λαβία οπότε ως πρόεδρος θα σας παρουσιάσω τις προτάσεις του εισηγητή μας. Λοιπόν, έχετε εκεί στο περιοδικό μας με τα νέα την παρουσίαση. Το 12 και το 15 αντιστοιχούν σε θέματα κινητικότητας ε, σε σχέση με το Ταμείο Προσαρμογής στην ε, Παγκοσμιοποίηση, δηλαδή οι πιστώσεις που μεταφέρονται σε αυτό το κονδύλι. Σας προτείνω ε, μία ενιαία ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της μεταφοράς, κατά, αποχές. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Η ίδια ψήφος ο ίδιος συσχετισμός. Άρα 12 και 15 εγκρίνονται. Τώρα, ως προς την μεταφορά υπαριθμών 20, πρόκειται για ένα αποθεματικό του 13, αναμένοντας επαρκείς ε, πληροφορίες. Ίσως υπάρχουν στο μεταξύ και έχουν δοθεί στον εισηγητή. Πρόκειται για μια μεταφορά 12 ευρώ υποχρεώσεις και 7.150.000 για τις πληρωμές υπέρ. Κατά. Αρτόγκ. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα. Ε, υποβάλλουμε και τα υπόλοιπα σε ψηφοφορία. Τις υπόλοιπες θέσεις. Άρση άρση επιφύλαξη επί του αποθεματικού. Ωραία. Μπορούν να αρθούν οι επιφυλάξεις διότι πληρούνται οι όροι ως προς το αποθεματικό. 24 υπέρ. Επί του 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Επί του 25 υπέρ. Κατά. Αρτόγκ. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία για τα άλλα τμήματα. Ο συνάδελφος είναι εδώ και του δίνω το λόγο. Uh, thank you, I have uh, two... Ο κύριος Βον. Υπάρχουν δύο αιτήματα μεταφοράς. Με την άδειά σας θα τις δω από κοινού για να μην χάνουμε χρόνο. Η πρώτη αφορά το ελεγκτικό συνέδριο. Πρόκειται για μία μικρή μεταφορά 145.000 ευρώ. Το ελεγκτικό ε, έχει ορισμένα χρήματα διότι έχουν εγκαταλείψει ένα κτίριο και έτσι έχουν αποταμιευθεί ορισμένα εκατομμύρια τα οποία θα μεταφερθούν σε γραμμές του προϋπολογισμού ε, σε σχέση με την προσχώρηση της Κροατίας δηλαδή. Εκεί μεταφέρονται αυτά τα κονδύλια. Έτσι γίνεται η μεταφορά. Ως προς τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου θα θυμόσαστε ότι στον προϋπολογισμό υπάρχει στην ΙΜΑΣ ένα εκατομμύριο ευρώ που έχουν αποταμιευθεί και ζητούμε να αρθεί η αποταμίευση για πέντε πράγματα. Καταρχήν τη βελτίωση για τις διασκέψεις, ε, τις τηλεδιασκέψεις έτσι ώστε να ε, αποταμιεύσουμε και να εξοικονομήσουμε. Επίσης, ε, catering για τη βελτίωση αυτής της υπηρεσίας, εφοδιασμού, εστίασης, τρίτον, ε, διαχείριση αποβλήτων, οικολογικών αποβλήτων, προβλέπονται διάφορα, διάφοροι χώροι γι' αυτό στους τόπους εργασίας, επίσης ηλεκτρικά οχήματα για τη μεταφορά ε, αγαθών για αποταμίευση και πάλι και εξοικονόμηση, με συγχωρείτε, και επίσης αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων για το προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και για τα μέλη αν το επιθυμούν. Αυτές είναι οι πέντε γραμμές του υπερεπολίσμού για, τα, για το ένα εκατομμύριο της μεταφοράς αυτής. Εκεί θα απορροφηθούν και σας παρακαλώ να δεχτείτε αυτή τη μεταφορά αυτή την απορρόφηση. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ωραία. Ηλεκτρικά ποδήλατα για τα μέλη και ε, κανονικά για το προσωπικό. Κύριε Αρτών, τι λέτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω ένα μικρό σημείο από πλευράς ε, ελεκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά το VIB 06C 13 θεωρώ ότι είναι πολύ εντυπωσιακό ότι παρενοχλείται η Επιτροπή Προπολογισμών για 10.000 ευρώ επιπλέον για την αύξηση αριθμού καφέδων που ζητήθηκαν. Τι... Αυτό ήθελα να επισημάνω. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν αφορά τον καφέ αποκλειστικά. Γενικά ίσως και ποτά που προσδίδουν μεγαλύτερη ενέργεια. Boosters. Εισηγητής. Ε, είναι ένα μικρό μέρος της ε, μεταφοράς. Ε, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, άρα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, φωτοτυπικά, συμβάσεις για τα φωτοτυπικά. Γι' αυτό μιλάμε και για ποτά μετά από ένα θερμό καλοκαίρι. Δεν ξέρω κατά πόσο τα 10.000 ευρώ αιτιολογούνται. Εν πάση περιπτώσει πρόκειται για διαβούλευση. Είναι τεχνικής υφής αυτή η μεταφορά, δεν μπορούμε να αντιταχθούμε, διότι πρόκειται για ένα μελιτέο ποσό. Ο κύριος Αρτόγκ έχει δίκιο. Θα πρέπει να προσέξουμε τη διατύπωση ως προς τις αιτήσει μεταφοράς. Ωραία. Μεταφορές του ελεγκτικού που ζητήθηκαν από το ελεγκτικό. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Τρεις αποχές εγκρίνεται η μεταφορά. Ως προς το κοινοβούλιο υπέρ. Υπέρ της μεταφοράς για τα ποδήλατα. Κατά. Ένας. Αποχές εγκρίνεται λάβαμε και ένα άλλο αίτημα μεταφοράς από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, αλλά σε μία γλώσσα μόνο. Είμαι ο μόνος που γνωρίζει αυτή τη γλώσσα. Άρα δεν πληρούνται οι όροι από νομικής πλευράς για να γίνει ψηφοφορία, άρα θα ψηφίσουμε την επόμενη φορά. Ως προς την πολιτική κατασκευών, η Μόνικα Χολμάιερ, Buildings Policy, την άλλη φορά θα μας ε, θα το ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Euh, Άρα έληξαν οι ψηφοφορίες. Alors, je euh, euh, Θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στη νομική υπηρεσία, στο νομικό σύμβουλο που βρίσκεται. Ο κύριος Πενέρα, εδώ είναι, μαζί μας. Δεν είμαι συνηθισμένος στην μεγάλη αυτή αίθουσα, την οποία χρησιμοποιούμε συνήθως για τριμερείς διαλόγους. Δεν είμαι συνηθισμένος. Είσαστε κομιστής μιας καλής είδησης, την οποία και θα μας ε, εξηγείτε. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να σχολιάσω αυτή τη σημαντική απόφαση. Πρόκειται για μία σειρά ζητημάτων του προϋπολογισμού που ξεχνάμε. Η πρώτη διαφορά αφορά ζητήματα του προϋπολογισμού. Ήδη το 79 είχαν γίνει οι πρώτες προσφυγές μετά το 82-83 και είχαμε τη μεγάλη απόφαση του 86 μετά είχαμε την απόφαση για το Συμβούλιο και τα, την ε, μεταχείριση των υπολείπων του προϋπολογισμού, μια άλλη απόφαση το 1995 και μια άλλη σημαντική απόφαση τώρα, διότι θα ορίσει την κατάσταση μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μπορώ να σας πω ότι η απόφαση αυτή είναι βανάγνωστη, θα σας δώσω μια συνοπτική εικόνα της απόφασης. Πρώτον, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ε, είναι η μόνη αρχή που μπορεί να αποφασίσει το, επί του προϋπολογισμού. Από, από πού ανακύπτει η διαφορά. Η συνθήκη του Λουξεμβούργου του Απριλίου 1970 όριζε τον πρόεδρο του Συμβουλίου για να υπογράψει για τον προπολογισμό. Από το 1975 ορίζεται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου για να αποφασίσει. Το Συμβούλιο αμφισβητεί αυτά τα δεδομένα. Το Συμβούλιο κρίνει ξεπερασμένη αυτή την απόφαση θα σας διαβάσω λοιπόν την απόφαση της 3ης Ιουλίου του 86 και αναφέρω, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θεωρεί ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού ε, έχει ολοκληρωθεί με την υπογραφή του προϋπολογισμού γι' αυτό. Ο προϋπολογισμός ε, θεωρείται οριστικός προς τα τρία θεσμικά όργανα και έτσι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου με αυτή την πράξη δυνάμει μιας διαδικασίας με βάση την κοινή δράση των τριών θεσμικών οργάνων υπογράφει αυτή την πράξη όχι χωριστά, αλλά ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο θεωρούσε ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουν αλλάξει τα πράγματα και η δημοσιονομική διαδικασία είναι διαφορετική. Εφόσον πρόκειται για μια διαδικασία πρωτοβουλίας, τότε θα έπρεπε να νομοθετήσει κάποιος και να υπογράψει κάποιος. Ε, δεν ήταν σαφές για το Συμβούλιο ότι κλείνει τη διαδικασία του προϋπολογισμού το Κοινοβούλιο και θεωρούσε ότι τόσο ο πρόεδρος του Συμβουλίου όσο και του Κοινοβουλίου πρέπει να προσυπογράψουν, να υπογράψουν αυτή την πράξη. Δυνάμει του άρθρου 314 παράγραφος 10 όπου ο πρόεδρος ε, αποφαίνεται για τον προϋπολογισμό ε, αυτό ακριβώς αμφισβητούσε το Συμβούλιο. Το δικαστήριο πώς αποφάνθηκε. Θεωρεί ότι η διαδικασία του προπολογισμού δεν αφορά την κοινή υπογραφή της πράξης από τους δύο πρόεδρους. Δυνάμει του άρθρου 314, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου διαπιστώνει μετά από την επαλήθευση της ε, διαδικασίας ότι εγκρίνεται οριστικά ο προϋπολογισμός δυνάμει της διαδικασίας, ε, της οριστικής αυτής διαδικασίας, η οποία τίθεται ενισχύει βασιζόμαστε στο άρθρο 203 της ε, προγενέστερης συνθήκης και νυν άρθρο 314. Η πράξη αυτή υπογράφεται από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου που λαμβάνει την οριστική απόφαση. Άρα ο προϋπολογισμός τίθεται εν ισχύ, έχει υποχρεωτική ισχύ. Αυτή ήταν η απόφαση του 86 που είχε ληφθεί από το δικαστήριο το 86. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκε αυτό το πλαίσιο, όχι με χρονολογική σειρά, από, την, ε, από το πεδίο εφαρμογής αυτής της δράσης. Τι κάνει ο πρόεδρος μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Αυτά που σας διάβασα ήταν οι παράγραφοι 50 και 51 της απόφασης. Τώρα θα σας διαβάσω τις παραγράφους 66 και 67. Συνάπτεται συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό. Το γεγονός ότι τα δύο αυτά θεσμικά όργανα είχαν εκφράσει διαφορά για την τυποποίηση αυτής της απόφασης δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος της 15 ε, ε, Δεκεμβρίου 2010 δεν θεώρησε ότι εγκρίνεται οριστικά αυτός ο προϋπολογισμός και συνεπώς μόνο ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου μπορεί να υπογράψει αυτή την πράξη και άρα δεν τίθεται θέμα παραβίασης του ε, ρυθμιστικού αυτού πλαισίου. Έτσι τηρούμε τη διαδικασία του προϋπολογισμού. μπορούμε να αντλήσουμε ένα δίδαγμα ως προς τη φύση του προϋπολογισμού. Τι σημαίνει η οριστική πράξη περί προϋπολογισμού. Ήδη το 86 είχαμε όλα τα στοιχεία και το 95 στη συνέχεια. Ο προϋπολογισμός δεν είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Είναι ένα λογιστικό έγγραφο. Η μόνη νομοθετική πράξη είναι η πράξη που υπογράφει ο πρόεδρος θα μπορούσαμε να δώσουμε, να αναφερθούμε στο εξής συμπέρασμα. Αλλά πριν θα ήθελα να σας αναφέρω τη συλλογιστική του δικαστηρίου. Η, το άρθρο 314 μιλά για μία ειδική νομοθετική πράξη. Πρόκειται όμως για ένα λογιστικό έγγραφο με τις εκτιμήσεις και προβλέψεις δαπανών. Αυτό το έγγραφο, σε αυτό το έγγραφο υπάρχει ένα παράρτημα μετά από την επαλήθευση της διαδικασίας αυτής, βασιζόμαστε στο άρθρο 314 για την οριστική αυτή πράξη, δηλαδή την έγκριση του προϋπολογισμού. Ακόμα και αν βασιζόμαστε λοιπόν σε μια ειδική νομοθετική διαδικασία, η πράξη αυτή εξαιτία της φύσης του προπολογισμού θεωρείται, δεν θεωρείται νομοθετική πράξη δύναμη του άρθρου 314 αποτελεί μία πράξη που μπορεί να προσβληθεί δύναμη του άρθρου 263. Άρα δεν πρόκειται για νομοθετική πράξη, αλλά νομική, που ελέγχεται από το δικαστήριο. Αυτά όλα σας τα λέω, διότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ποια νομικά κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να κρίνουμε την λυσιτέλεια ενός ε, ε, νομικού εγγράφου, με συγχωρείτε, ενός λογιστικού εγγράφου. Δεν ξέρω κατά πόσο το δικαστήριο ήθελε να κρίνει την εμβέλεια αυτών των πράξεων, αλλά, εν περιπτώσει, αυτό είναι το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης και αυτό ήθελα να υπογραμμίσω ενώπιόν σας. Έτσι βάλαμε τα πράγματα σε μία τάξη. Το, το Συμβούλιο δεν ήθελε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, αυτή η διαφορά. Πρόκειται για μία πύρια νίκη όμως. Γιατί αν είχαμε να κάνουμε με μία απόφαση που θεωρούσε ότι ο πρόεδρος ε, δεν έχει την αρμοδιότητα να υπογράψει αυτή την πράξη που έχει εκτελεστική ισχύ, αλλά μπορούσε ή θα έπρεπε να γίνει κοινή υπογραφή και έγκριση από τους δύο Προέδρους, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, θα ήταν πολύ αρνητικό. Πρόκειται για μία σχηνοτενή διαδικασία που έχει αρχίσει το 1995. Τώρα, οι τροποποιήσεις με τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι συγκεκριμένες. Ορισμένα στοιχεία δεν έχουν μεταφερθεί σωστά και γι' αυτό υπάρχουν, ε, υπάρχει μία έλλειψη ισορροπίας με βάση την τακτική νομοθετική διαδικασία ή την ειδική διαδικασία νομοθέτησης. Πολλές φορές όταν τα αναλύουμε όλα αυτά, μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τύπου συμβουλίου. πάση περιπτώσει τα νέα είναι πολύ καλά για μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Ρικάρντο Πάσος και τον, τον κύριο Γκάουτσι, ο οποίος τώρα βρίσκεται ε, πλαισιών της ε, νομικές υπηρεσίες της ε, Κομισιόν. Η νομική υπηρεσία το 2009 είχαμε κοινοποιήσει στον πρόεδρο ότι δεν έπρεπε να επιτρέψει τη λανθασμένη αυτή η ερμηνεία του Συμβουλίου και τώρα επιβεβαιώθηκε η θέση μας. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Merci, cher ami. Ευχαριστώ αγαπητέ φίλε. Νομίζω ότι είναι χαρμόσυνη η είδηση. Είναι ουσιώδης νίκη. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικονομικής βάσης, ε, μάχης που δεκαετίες τώρα διεξάγεται από το Κοινοβουλίο μας και από πλευρά της Επιτροπής Πρεπολισμών. Αγαπητέ φίλε, θέλω να σας συγχαρώ και όλους σας τους συνεργάτες, διότι επιτύχατε ε, ε, να πείσετε με την επιχειρηματολογία σας το δικαστήριο. Γιατί είχαμε καταλήξει σε μια κατάσταση που ήταν ε, από ορισμένε απόψει γελία. Πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Συμβούλιο, η Προεδρία του Συμβουλίου, άφηνε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου στο τέλος της ψηφοφορίας ε, στην Ολομέλεια να υπογράψει τον προπολογισμό. Αυτό μας επέτρεπε μετά τη λήξη των ε, ψηφοφοριών να έχουμε στην Ολομέλεια μία οικογενειακή φωτογραφία, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, πλαισιωμένος από τον πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμών, τους εισηγητές, τον επίτροπο επί του προϋπολογισμού και ενδεχομένως ε, σε μία θεσούλα στην άκρη βάζαμε και τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Μετά την ε, έναρξη ισχύω της συνθήκης Λισαβόνας περάσαμε σε μία γραφική κατάσταση όπου το σχέδιο προπολογισμού ε, το βάζαμε από κάτω από τα έδρα, από το θεωρία του Προεδρείου και μετά τρέχανε ο πρόεδρος του Συμβουλίου και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου για το ποιος θα υπογράψει πρώτος. Και δεν υπήρχε καμιά φωτογραφία μετά. Τώρα η κατάσταση είναι πολύ πιο αξιοπρεπής, ε, πολύ σύμφωνη με το πνεύμα των συνθήκων και που ε, ε, είναι σκόπιμη και για το Κοινοβούλιο. Ο Ζωάν Ντεάν μου είπε επίσης ότι εφόσον το δικαστήριο είναι τη σοφία του κάνει μια αρκετά αναπάντεχη ανάλυση αλλά η απόφασή του είναι κυρίαρχη όπου θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα απλώς λογιστικό έγγραφο και ότι η νομοθετική πράξη είναι η υπογραφή του Προέδρου. Αν αυτή λοιπόν είναι η νομική ερμηνεία ε, των συνθήκων που ισχύει, το Κοινοβούλιο έχει ένα ιδιαίτερα βάσιμο επιχείρημα για να ισχυριστεί, να θεωρήσει ότι κατά κανένα τρόπο, ούτε νομικά ούτε πολιτικά, η ε, παρούσα πρακτική του Συμβουλίου των Υπουργών, με βάση την οποία το Συμβούλιο αποστέλει στα Εθνικά Κοινοβούλια το σχέδιο προπλησμού της Επιτροπής και τους δίνει 8 εβδομάδες για να υποβάλουν ενδεχομένω ε, τη γνώμη τους για την ε, ε, συμβατότητά του με βάση το πρωτόκολλο 2 με την αρχή της επικορικότητας και τις συνθήκες. Δεν ξέρω αν επ' αυτού θέλει ο νομικός μας σύμβουλος να μας δώσει τη γνώμη του το πρωτοκόλλο 1 και το πρωτόκολλο 2, εδώ πρόκειται για το πρωτόκολλο 1, μιλάει για σχέδια νομοθετικών πράξεων. Με τη στενή έννοια, στρίκτο ένσου, μας είπαν ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι νομοθετική πράξη. Ότι η νομοθετική πράξη είναι αυτή που διαπιστώνει ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, λέει ο Νομικός Συμβουλός. Από την άλλη μεριά, δεν χρειάζεται να επιμένουμε ιδιαίτερα στις κακές πρακτικές του ε, Συμβουλίου γιατί ε, επιβάλλεται από τις προθεσμίες που προβλέπει το άρθρο 314 1η Ιουλίου κτλ. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, θα είναι δύσκολο να επιβάλλουμε στο Συμβούλιο ή ε, ουδήποτε τύπου πειθαρχία γιατί πάνω κάτω κάνει ό,τι θέλει. Δεν πρόκειται για μια πράξη που μας βλάπτει. Οπότε βεβαίω είναι κακή συνήθεια, αλλά όσο δεν παραβιάζει τις υποχρεωτικές ε, ε, ρήτρες του άρθρου 314 δεν μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα πιστεί από αυτήν την απόφαση του δικαστηρίου που φυσικά ε, δεν του είναι αρεστή. Πρόεδρος. Εντάξει, στην πράξη το Συμβούλιο, όπως και εμείς, ε, πρέπει να ε, σεβαστεί πολύ συγκεκριμένες ε, προθεσμίες για την έγκριση του προπολογισμού. Λόγω αυτού του χρονοδιαγράμματος, όπως διαπιστώσαμε από τότε που ισχύει η Συνθήκη της Λισαβόνας, κάθε χρόνο, στην πράξη, το σχέδιο προπολογισμού δεν το ψηφίζει το Συμβούλιο των Υπουργών Προπολογισμού. Είναι γραπτή διαδικασία. Γιατί οκτώ εβδομάδε σημαίνει ότι είμαστε στον Αύγουστο, δεν συνεδριάζουν οι Υπουργοί Προπολογισμών και πολλέ φορέ δεν έρχονται καν στι Βρυξέλλε. Γενικώ, άρα πολύ λιγότερο θα έρθουν τον Αύγουστο. Ούτε καν οι πρέσβει. Είναι μια είδου ε, γραπτή διαδικασία. Και τελικά το σχέδιο προπολογισμού της Ένωσης δεν ε, διαμορφώνεται μετά από μια πραγματική πολιτική δημόσια συζήτηση στο επίπεδο του Συμβουλίου των Υπουργών. Αλλά έχετε δίκιο δεν είναι κυρίως ε, νομικό, είναι κυρίως ε, πολιτικό θέμα ουσίας. Το τονίσαμε την πρώτη χρονιά ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι μια μάχη ε, που δεν έχουμε ακόμη κερδίσει. Θα το επιχειρήσουμε. Η διάδοχή μας δηλαδή. Λοιπόν, ωραία κερδίσαμε από νομική πλευρά. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου υπογράφει τον προπολογισμό, εμείς και οι βουλευτές και κυρίως η Επιτροπή Προπολογισμών πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει, ούτως ώστε ε, τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται ε, στον προπολογισμό να είναι αυτά που εμείς επιθυμούμε και όχι αυτά που επιθυμεί το Συμβούλιο. Εδώ είναι η πολιτική συζήτηση γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, και κάποιο παζάρι, να υπογράφουν εκείνοι και εμείς να βάζουμε τις πιστώσεις που θέλουμε. Ευχαριστώ τον ε, νομικό μας σύμβουλο, τον συγχαίρω. Μας μένουν ορισμένα ε, ακόμη σημεία, αλλά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αρκετά γρήγορα. Για τις πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές και την διοργανική συμφωνία. Δεν ξέρω εάν ο Ζαν έχει να μας πει τίποτα. Α, Δεν χρειάζεται μεγάλη συζήτηση, ε, μακροσκελή συζήτηση. Ε, κάνουμε ενημέρωση για το τι συμβαίνει. Δεν έχει συμβεί τίποτα από την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, που είχαμε Ολομέλεια δηλαδή, θα θυμάστε, ότι εγκρίναμε στην Ολομέλεια το DAB αριθμός 2, σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2013 και ο Πρόεδρος αποφάσισε η τελική ψηφοφορία για την νομική πλευρά των ε, δημοσιονομικών προοπτικών, δηλαδή τον κανονισμό για τις πολιτικές προοπτικές, τη Οργανική Συμφωνία και την απόφαση για τους ίδιους πόρους, για την οποία απλώ ε, ε, μας διαβουλεύονται. Ο πρόεδρος μπορεί να λοιπόν αποφάσει όλα αυτά, η ψηφοφορία, η τελική για όλα αυτά, να αναβληθεί για τον Οκτώβριο. Ζητήσαμε μια νέα προθεσμία από την ΑΦΚΟ του είπαμε δηλαδή να αναβάλουν και εκείνοι την ψηφοφορία τους από αυτού. Πήγα εγώ ίδιος ε, προχθές στην ΑΦΚΟ. Η ΑΦΚΟ εκπονεί μία έκθεση που περιέχει ε, αυτολεξή τις ε, συστάσεις που τους είχαμε αποστείλει, να εργαζόμαστε άρεστα. Σήμερα το πρωί ε, εξετάσαμε την κατάσταση όσον αφορά τις πληρωμές ευευκαιρία τη συζήτηση για το σχέδιο προπολογισμού του 2014 και εκτός αν κάποιοι από εσά ε, έχουν σχόλια ε, να περιοριστούμε σε αυτά και φυσικά ήδη από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει ακόμη ενημέρωση. Την επόμενη εβδομάδα και να δούμε πώς θα ε, κατανείμουμε τα καθήκοντά μας. Στις 26 έχουμε το απόγευμα την Επιτροπή Προπολισμών και το πρωί συντονιστές κατόπιν δύο η ώρα ε, την συνάντηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τις πληρωμές και η συνεδρίαση η δική μας θα αρχίσει στις 3 και 30. Έχετε σχόλια? Ωραία. Α, έχετε. Α, παρακαλώ. Έλγα, έχετε μια ερώτηση. Τι ώρα η συνεδρίαση των συντονιστών? 10 και 30. Θα το επιβεβαιώσουμε. 10 και 30, 12 και 30 είναι σημαντική συνεδρίαση. Γιατί είναι τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών πριν από την ψήφιση των τροπολογιών που θα γίνει 2 και 3 Οκτωβρίου. Άλλε ερωτήσει, παρακαλώ. Κύριο Μπεκμανή. Επειδή μιλάμε για αυτές τις πολιτικές προοπτικές, να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής Προπολογισμών στην επιστολή που στείλαμε στην αρχή της συνεδρίασης ε, για να δώσουμε συνέχιση, γιατί γι' αυτό αναβάλαμε την ε, ψηφοφορία, είναι ότι γιατί επειδή υπάρχουν ε, διαφορές για δύο βασικούς κανονισμούς, συνοχή και άγκρη. Δεν ξέρω τι γίνεται με την άγκρη, αλλά για τη συνοχή Έχουμε, είχαμε πάνω από 70 τριμερείς διαλόγους. Σήμερα έγινε ο τελευταίος και θα γίνει ο επόμενος την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν θα επιτύχουμε συμβασμούς για δύο θέματα με το Συμβούλιο. Ο ένας είναι το αποθεματικό για την ε, απόδοση και το δεύτερο είναι αιρεσιμότητα. Ιδίως αυτό το θέμα αιρεσιμότητα. Για το δεύτερο αυτό θέμα το Κοινοβούλιο απέχει πολύ από το Συμβούλιο, δεν υπάρχει ενδεχόμενο ε, συμβασμού και το είπαν και οι δύο. Τι θα γίνει λοιπόν με την ψηφοφορία για τι πολιτικέ προοπτικέ, τι θέλουμε να κάνει η Επιτροπή Προπολογισμών, εάν εξακολουθήσει η ίδια κατάσταση, εάν δηλαδή δεν καταλήξουμε σε συμβασμό για έναν ή και για του δύο αυτού του συμβασμού. Ο διάλογο ε, για την ε, συνοχή δεν αλλάζει βέβαια τα αριθμητικά στοιχεία Υπάρχει συμφωνία μεταξύ Κομισιόν και Συμβουλίου. Αλλά ε, σε αυτή την επιστολή το αναφέρουμε ως εμπόδιο. Ήθελα να σε ενημερώσω ότι δεν υπάρχει λοιπόν προοπτική συμφωνία. Τι θα κάνουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε είναι πολιτικό θέμα θεμελιώδη σημασία. Απάντηση. Περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία. Αν εξακολουθήσουν να υπάρχουν πολιτικές δυσχέρειες σε, για πρωταρχικά θέματα, αν είναι δευτερεύοντα θέματα, δεν πειράζει και τόσο πολύ, αλλά αυτά είναι πρωτεύοντα. Δεν ξέρω εάν υπάρχουν κάποια άλλα μέλη της Αγκρή, ο Λαβία Λύπη, αλλά και αυτοί έχουν τρία-τέσσερα λοιπόν σημαντικά θέματα όπου υπάρχουν δυσχέρειες. Ελπίζουμε λοιπόν οι προθεσμίες της Τετάρτης 2 Οκτωβρίου, η προθεσμία της 2 Οκτωβρίου να είναι αρκετά εντυπωσιακή για τους συμμετέχοντες στους διαλόγους για να επιτύχουν μέχρι τότε συμβιβασμό. Ο πρόεδρος Σούλτς γνωρίζει πολύ καλά τις δυσχέρειες του εγχειρήματο και είπε ότι είναι διατεθειμένος να προτείνει στον πρόεδρο Μπαρόζο και τη Λιθουανική Προεδρία να υπάρξει άλλη μία συνάντηση κορυφής των Προέδρων των Τριών Θεσμικών Οργάνων για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο με βάση τη ε, διαδικασία του άρθρου 324 της Συνθήκης για την Ένωση ε, την οποία ε, διαδικασία αξιοποιήσαμε και για να επιτύχουμε συμφωνία για τις πολιτικές προοπτικές. Για τα δύο σημεία που αναφέρατε για το Ταμείο Συνοχής. Για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Όπως λέτε, από πλευράς αρχής είμαστε αντιδιαμετρικά ε, αντίθετοι με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Αλλά για το άλλο θέμα δεν είμαι και τόσο ανήσυχος γιατί παρά τα φαινόμενα φαίνεται, διαφαίνεται τελικό συμβασμός. Αλλά τονίζω ότι για το αποθεματικό αποδοτικότητας, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι οι διαφορές μεταξύ 7 και 5% ε, έχουν επίπτωση στις πιστώσεις πληρωμών. Οπότε, το Συμβούλιο αλλά και η Επιτροπή θεωρούν ότι τίθεται να αμφιβόλω το ανώτατο όριο πληρωμών. Αναμφίβολα λοιπόν πρέπει οι διαπραγματευτές μας να το εξετάσουν με μεγάλη προσοχή. Να δούμε δηλαδή τι τμήματα του Ταμείου Συνοχής θα μπουν ε, στο αποθεματικό για να ενθαρρύνουμε την αποδοτικότητα και την σωστή διαχείριση, αλλά τι επιπτώσεις από την άλλη μεριά έχει αυτό το ανώτατο όριο πληρωμών. Μπορούμε να βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε χωρί να φυγεί το ανώτατο όριο πληρωμών. Οι πληροφορίε που έχω. Με οθούν στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι πιο δυσχερέ θέμα από την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Αλλά βέβαια εσεί διαπραγματεύεστε, εσεί είστε αρμόδιο. Αλλά εάν αντίθετα με την αισιοδοξία που εκφράζω δεν υπάρξει λύση, δεν καταλήξετε σε συμβασμό που να θεωρείται αποδεκτό, τότε η θέση της διάσκεψης των Προέδρων είναι ότι θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε, εφόσον τα θέματα αυτά είναι πρωταρχικά, θα περιμένουμε το Συμβούλιο να κάνει τις αναγκαίες υποχωρήσεις. Μια πρώτη ενέργεια είναι να αναβάλουμε ε, κατά ένα μήνα, κατά δύο ολομέλειες, μέχρι τη δεύτερη του Οκτωβρίου την τελική ψηφοφορία με αυτές τις δύο απαιτήσει που ήδη αναφέρατε. Θα δούμε μέχρι τη δεύτερη ολομέλεια του ε, Οκτωβρίου αν θα έχει σημειωθεί πρόοδος. Ε, αν δεν έχουμε τα επιπλέον 3,9 δις θα περιμένουμε μέχρι να τα λάβουμε αν υπάρχουν ακόμη από πλευρά μα ε, θεμελιώδει πολιτικέ αντιρρήσει όπω αυτέ που αναφέρετε για την πολιτική βάση, για την νομική συγγνώμη βάση, θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο περισσότερο. Είμαι πεπισμένο ότι ο πρόεδρο Σούλτ θα τα συζητήσει την επόμενη φορά που θα συναντηθεί με τι πολιτικέ ομάδε και φυσικά θα υποβάλει στη διάσκεψη των Προέδρων πρόταση απόφαση που θα προβλέπεται αυτή η δυνατότητα. Πολύ σύντομα νομίζω θα συμβεί αυτό. Στι επόμενε δύο-τρει εβδομάδε με βάση τι θα συμβεί και στον επόμενο τριμερή διάλογο. Θα ε, εξετάσει λοιπόν το ενδεχόμενο συνάντηση κορυφή των τριών προέδρων των θεσμών. Ευχαριστώ. Άλλα θέματα. Έχουμε το σημείο 11, το σημείο 11 γιατί τα άλλα τα έχουμε ε, αναβάλει, δηλαδή η εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες σε επενδυτικά έργα εκτός Ένωσης. Ο Ιβάιλο δεν είναι εδώ, αλλά ο Γκέρεν θα τον αντικαταστήσει. Ναι, είχα υποσχεθεί να μιλήσω για αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά τα σύνορα Βουλγαρίας, Τουρκίας και Ελλάδας. Ε, ε, εκεί θα πρέπει να εξετάσουμε κάποια ενδιαφέροντα σημεία. Πρόκειται για την εντολή την εξωτερική της ε, στην ΕΤΕΠ. Θα θυμάστε ότι είχαμε πριν από κάποια χρόνια ένα τέτοιο θέμα παρόμοιο στην ατζέντα. Τότε αναθεωρήθηκε η εντολή. Τώρα συζητάμε την εντολή την καινούργια μετά το 2013 για τη νέα δημοσιονομική προοπτική. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχε ε, δανείσει χρήματα εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε με ίδιο κίνδυνο ως ξεχωριστή τράπεζα ή με ασφάλεια του κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η όλη ιδέα σε ό,τι αφορά αυτόν τον εξωτερικό δανεισμό ήταν ασφαλώς ότι επρόκειτο για ένα μέσο της Ένωσης για να πετύχει εξωτερικούς στόχους και δεσμεύσεις, δίδοντας πόρους ε, μέσω αυτού της διαδικασίας δανεισμού της Τράπεζας Επενδύσεως. Οι ασφαλίσεις ασφαλίζονται με, από ένα ταμείο που συμπληρώνεται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και ε, η έκταση των εγγύσεων καθορίζονται από την ΕΤΕΠ. Και γι' αυτό λοιπόν η απόφαση που αυτό να πάρουμε είναι πολύ σημαντική. Η ιδέα είναι ότι το μοντέλο αυτό ε, δουλεύει σε όλε τι περιφέρειε τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στα κράτη-μέλη εκείνη, αλλά και σε ενδεχόμενα κράτη-μέλη, στα Βαλκάνια, στι ε, γειτονικέ χώρε, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και στην Αφρική υπάρχει ξεχωριστή εντολή. Όπως σας, λέω, όπως σας είπα, ε, πλέον αυτή η εντολή θα έχει προθεσμία μέχρι και φέτος. Άρα σύντομα θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα γίνει από το 2014 και εξή. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει συνολική εντολή 28 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα δεν μιλάμε για εκατομμύρια, μιλάμε για δισεκατομμύρια και μάλιστα για πολλά. Και αυτό σε δύο τμήματα 25 εκατομμύρια, ε, δισεκατομμύρια έχουμε ε, ως ανώτατο όριο και υπάρχει πρόταση να προσθεθούν άλλα 3 δισεκατομμύρια. Αυτό μέχρι την 1,5 αναθεώρηση του 2017. Το πρόβλημα είναι, θεωρεί ο εισηγητής, ότι το όριο αυτό ουσιαστικά αποτελεί μία περικοπή, μείωση σε σχέση με τα τρέχουσα άνωτα τα όρια 30 σχεδόν ε, δισεκατομμύρια, 29 και μισό. Τώρα μιλάμε για μείωση δηλαδή στα 28 δισεκατομμύρια, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Μιλάμε για πολλά χρήματα και γι' αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Η μείωση δε θα πλήξει σχεδόν όλες τις περιοχές, ιδιαίτερως στην Λατινική Αμερική και την ε, Νότιο Αφρική. Ο εισηγητής παρουσίασε ένα σχέδιο έκθεσης 40 τροπολογίε κατατέθηκαν και κάποια θέματα θα ήθελα να τα, θα ήθελα να τα τονίσει. Τα αριθμητικά στοιχεία, τα θέματα διαφάνεια σε σχέση με του εμπλεκόμενου φορεί και την καλύτερη εναρμόνιση με τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και το καθεξής. Σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία, προτείνει να επανέλθει το ισχύον άνατατο όριο και να υπάρξει αύξηση δηλαδή σε ό,τι αφορά το βασικό ποσό κατά ένα εκατομμύριο και σε ό,τι αφορά τα ε, ενδεχόμενα προσθήκη. Να πάμε δηλαδή στα 30 δισεκατομμύρια. Το βασικό επιχείρημα υπέρ ε, αυτού είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μέσω της EIB ε, επενδύσεις με πολύ μεγάλη αποδοτικότητα, μεγάλη μόχλευση και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το, ο αντίκτυπος των δύο επιπλέον δισεκατομμυρίων θα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Στο δεύτερο τμήμα των τροπολογιών του τώρα μιλά για θέματα διαφάνειας, ε, επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς και ούτω καθεξής, όπου θεωρεί ότι χρειάζεται βελτίωση σημαντικές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τους τοπικούς φορείς, αλλά και σε ό,τι αφορά την καλύτερη υποβολή εκθέσεων και αναφορών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις καλύτερες σχέσεις με τους εξωτερικούς χρηματοδότες. Αυτό λοιπόν αφορά το δεύτερο τμήμα των τροπολογιών. το τρίτο τμήμα των τροπολογιών τώρα. Αναφορικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον αντίκτυπό τους. Ο εισηγητής θεωρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξει κατά βάση τα ίδια στοιχεία τα οποία ανέφερε και στις προτάσεις της ενδιάμεσης αναθεώρησης του 2011. Ασφαλώς ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να είναι πολύ σόφρον σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές πολιτικές. τραπεζικές πολιτικές. Θα πρέπει παρόλα αυτά να διατηρηθούν αυτές οι υψηλές ε, αξιολογήσεις ό,τι αφορά την υποστοληπτική ικανότητα. Ωστόσο, ο δανεισμό θα πρέπει να συνάδει και με τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ο εισηγητή θεωρεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση, για παράδειγμα πολιτικέ όπω η αλλαγή του κλίματο, κοινωνικά πρότυπα, πρότυπα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποφυγή, φροντιαφυγή. Υπάρχουν διάφορε πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με τι οποίε θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση σε ό,τι αφορά τον δανεισμό αυτό. Αυτά λοιπόν ως προς την ουσία των προτάσεων. Αυτά ως παρουσίαση. Καλώς ορίζουμε προτάσεις και στις 26 Σεπτεμβρίου την άλλη εβδομάδα θα γίνει η ανταλλαγή απόψεων. 1η Οκτωβρίου θα είναι προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και στις 17 Οκτωβρίου θα ληφθεί η απόφαση, θα γίνει ψηφοφορία στα πλαίσια της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστούμε πολύ, Γκέραν. Υπάρχουν σχόλια ή ερωτήσεις ή Χέλγα. Ευχαριστώ, Γκέραν. Εκπροσωπώ τον... που εκπροσώπησε τον Ήβαλο. Τα πράγματα για μας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, οι προτάσεις δηλαδή. Θα επικεντρωθούμε σε κάποια συγκεκριμένα σημεία σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά θέματα ποσότητας. Θα θέλαμε να υπάρχει διαφορετική κατανομή. Θα θέλαμε να είναι 27 δισεκατομμύρια συν 3 σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα. Το αναφέρατε ήδη, αλλά θα θέλαμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη διατύπωση και σε, αν θέλετε στην αποφασιστικότητα ε, σε ό,τι αφορά την υποστήριξη πράσινων project, ε, ανανεώσιμες, βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως ε, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε πράσινο, στον πράσινο τομέα, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική το 2020 και τους σχετικούς στόχους που έχουν τεθεί. Και όπως λέμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, να επικεντρωθούμε στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και στις επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες για θέματα διαφάνειας τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι αιτήσεις εκθέσεις. Και θα ήταν ενδιαφέρον και σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση αναθεώρηση. Και εκεί να ρίξουμε μια δεύτερη ματιά στις δυνατότητες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό και σε θέματα κανονισμών περί διαφάνειας. Ύστερα θα θέλαμε να τονίσουμε θέματα του άρθρου 21 των συνθήκων σε ό,τι αφορά την πρόθεση της δημοκρατίας, των ανθρωπινών δικαιωμάτων, της βιώσιμης οικογενειακής ανάπτυξης και της ε, προώθησης των ευρωπαϊκών στόχων. Είναι κρίμα που το χρονοδιάγραμμα είναι τόσο αυστηρό. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην παρούσα φάση, άρα θα πρέπει αναγκαστικά να συνεργαστούμε πολύ στενά. Ευχαριστώ. Merci bien. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. Φαίνεται πως όχι, όπως υπενθύμησε και ο Γκέραν. Θα επεκταθούμε την επόμενη εβδομάδα με την παρουσία του Προέδρου της ΕΤΕ. Προβλέπεται ακρόαση στις 26, όπως ξέρετε. Άλλα σχόλια. Φαίνεται πως όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη, λύεται η συνεδρία, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.